Ο κύριος Νίκολσον. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συμφωνήσω με την έκφραση παράσταση προς τον γαλλικό λαό σήμερα το πρωί. Όλοι ε, αισθανόμαστε τι αισθάνονται. Οι τελευταίες εξελίξεις, η περαιτέρω παράταση της αβεβαιότητας, αναβολητικότητα δηλαδή, είναι αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, η παράταση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το πραγματικό πρόβλημα. Αλλά δεν θα εκπλαγείτε κύριε Μπαρνιέ γιατί εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα αυτό είναι το backstop. Δεν είχα αλλάξει άποψη από αυτού. Το backstop έχει δυσχεράνει τι διαπραγματεύσει από την αρχή και θα συνεχίσει να το κάνει όσο εμένετε στη θέση σα. Πρέπει να σα πω ότι η παράταση μέχρι τον Οκτώβριο δεν νομίζω ότι θα καταλήξει σε συμφωνία. Θεωρώ ότι θα χρειαστεί μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα νέο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να αλλάξουν απόψει. Θα πρέπει να δοθεί μια ε, νέα ευκαιρία για να απαντήσω αυτό το πρόβλημα. Κοιτάξτε, εάν είναι κανεί μέλο μια λέσχη, πρέπει να είναι πλήρε μέλο. Δεν μπορεί να είσαι μισό μέσα και μισό έξω. Και αυτό είναι το πρόβλημα με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν μου επιτρέπετε. Έχει φύγει ο κύριο Μπροκ, αλλά παρόλα αυτά θα είναι και η δική μου τελευταία ομιλία σε αυτό το σώμα μετά από 30 χρόνια. Και θέλω να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να σας πω ότι ήταν μεγάλη μου τιμή αλλά και χαρά να εκπροσωπήσω το λαό της Βόρειας σε αυτό το σώμα για 30 χρόνια. Τα πήγαμε καλά ορισμένε φορές και, μερικέ, και μερικές φορές ήταν ε, πολύ άσχημες οι καταστάσεις που αντιμετωπίσαμε όταν είχαμε και τρομοκρατικές επιθέσεις όπως εδώ. Και περάσαμε όλοι μέσα από αυτά. Αλλά στο σώμα αυτό ακούσαμε τον Ζακ Ντελόρ που εξέφρασε την αλληλεγγύη του με τον πληθυσμό της ε, Βόρειας Ιρλανδίας και όταν εγώ, ο Ιαν Πέισλι και ο Τζον Χιούμ πήγαμε να το δούμε, μας ρώτησε τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για σας και η Ευρώπη βοήθησε, έδωσε πάνω από δύο δις που βοήθησαν πολλούς ανθρώπους παντού στη Βόρεια Όπως είπα και εγώ, λοιπόν σας ε, αποχαιρετώ. Ελπίζω να συνεισέφερα εγώ πέρασα καλέ καταστάσει, ελπίζω να προσώπησα σωστά το λαό μου, γιατί είναι ένα περήφανο λαό, είναι ένα καταπληκτικό λαό, ο λαό τη Βόρεια Ιρλανδία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νίκολσον και επειδή έχουμε δουλέψει μαζί στην Επιτροπή Γεωργίας πρέπει να πω ότι όντως είχατε πολύ επικοδομητική στάση εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των εκλογέων σας εδώ και 30 χρόνια. Σε ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Νομίζαμε ότι η προηγούμενη ομιλία θα ήταν τελευταία, αλλά τελικά είχατε μια δυνατότητα ακόμη. Συγγνώμη που ε, δεν τηρώ το χρόνο τώρα. Και τώρα κύριε Άντερσον για λεπτό. Τίποτα δεν έχει αλλάξει το Λονδίνο παραβιάζει επιλεκτικά τι συμφωνίε τη Μεγάλη Παρασκευή. Το Δουβλίνο μα παραμελεί εμά στο βορρά. Άλλοι έξι μήνε αβεβαιότητας, διότι οι Βρετανοί αναβάλουν αυτά τα οποία συμφώνησαν ότι πρέπει να εφαρμόσουν το Δεκέμβριο του 2017. Το Brexit ε, αφαιρεί τα δικαιώματα του, του λαού συμπεριλαμβανόμενο και το δικαιώματο ψήφου, κάτι που ήταν ε, στην καρδιά του κινήματο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα πολιτικά δικαιώματα. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν εκλογέ που η συντηρητική και τον DUP δεν ήθελε και που τα δύο κόμματα τη ε, Νότια Ιρλανδία δεν ήθελαν να ψηφίσει ο Βορρά για αυτά. Α στείλουμε ένα σαφέ μήνυμα στο Λονδίνο, το Δουβλίνο και τι Βρυξέλλε. Α ε, επικρίνουμε το χάλι του Brexit αυτό τον πολιτικό βανδαλισμό. Όλοι οι ψηφοφόροι στην Ιρλανδία, εκλέγοντα ευρωβουλευτέ του Sinn μπορούν να κάνουν ένα βήμα προς την Ιρλανδική ενότητα που θα είναι ο δημοκρατικός τρόπος για να βγούμε από το Brexit. Θα είναι μια σωστή λογική απόφαση για να επιτύχουμε την Ιρλανδική ενότητα. Σας ευχαριστώ όλους. Έχει ζητηθεί μπλε κάρτα. Κύριε Κέλλη. Παρακαλώ. Κύριε Άντερσον, εσείς δέχεστε να σας διατυπώσει την ερώτηση ο κύριος Κέλλη. Κύριε Σκέλη, ξέρετε ότι δεν συνηθίζω να ρωτάω με μπλε κάρτα του συναδέλφου. Είναι η δεύτερη μου τα δέκα χρόνια που είμαι εδώ. Αλλά όταν μας λέει η κυρία Άντερσον ότι έχει καταληφθεί η υπόθεση της Βόρειας Ιρλανδίας και όταν ξέρουμε ότι με το backstop... Ένα λεπτό, ε, λέει η Πρόεδρος, κάντε την ερώτηση. Ναι, όταν όμως ε, δεν έρχονται να συμμετάσχουν σε κανένα κοινοβούλιο ή συνέλευση τα μέλη του κόμματός της, μα βλέπετε ότι εγώ είμαι εδώ κύριε Κέλλη. Το Σινφέιν ξεκάθαρα τοποθετήθηκε σε σχέση με την απόφαση της ε, Ιρλανδικής κυβέρνησης, η οποία είναι η μόνη η οποία στερεί το δικαίωμα της συμμετοχής στις ευρωεκλογές από τους υπηκόους της όταν δεν κατοικούν μέσα στην επικράτεια της Ιρλανδικής Δημοκρατίας. Το ξέρεις πολύ καλά, Τζον, όταν με τον Τζον Χιούμ πήγαν η μητέρα μου και ο πατέρας μου και όλοι οι συγγενείς μου στο Λονδίνο να αγωνιστούν με τα συλλαλητήρια ζητώντας ψήφο ισότιμη, δεν είχαν την εκπροσώπηση, δεν είχαν τη δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Τέλειωσε ο χρόνος σας. Κύριε Σμιθ, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ε, βεβαίως και είναι κάπως υπερβολικές όλες αυτές ε, οι δηλώσεις περί αποτυχίας και κατάρρευσης, αλλά θα ήθελα να πω, Πρόεδρε Τούσκ, όπως, λέει και ο, όπως έλεγε ο Τζον Λένον, μπορεί να είσαι ονειροπόλος, αλλά δεν είσαι ο μόνος. You're a dreamer, but you're not the only one. Ευχαριστώ λοιπόν για τις προσπάθειές σας, κύριε Τούσκ, και το χρόνο που αφιερώσατε για τη διέξοδο. Ε, ωστόσο, και ενώ των ευρωεκλογών, θέλω ένα μήνυμα να αποστείλω. Να αποκομίσουμε όλοι το δίδαγμα του Brexit, να το μάθουμε το μάθημα αυτό, γιατί το Brexit ε, καραδοκεί σε κάθε χώρα. Οι λαϊκιστές είναι επικίνδυνοι παντού και πρέπει να αποστείλουμε και θεωρώ ε, παρατηρητές στις εκλογές γιατί δεν θα είναι απαραίτητα καθαρή η εκλογική αναμέτρηση. Θα ήθελα να βεβαιωθούμε ότι θα γίνει γνήσια εκλογική αναμέτρηση και επίσης ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι μπορεί να προσπαθήσουν να εμποδίσουν την ανάδειξη καθαρού αποτελεσμού από τις εκλογές και αν το ξανακάνουν. Το κόμμα μου στην Σκοτία είναι έτοιμο για να γυρίσει στην Ευρώπη και θέλουμε να στηριζόμαστε σε εσά όπως μπορείτε και εσείς να στηρίζετε σε εμά. Η κυρία Γκέρλινγκ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εδώ παρισταμένους για την υπομονή, αλλά και την ηγετική στάση που επέδειξαν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, κύριε Τούσκ, ιδιαίτερος προς εσάς πρέπει να ε, ε, πω ευχαριστώ με όλα ε, στις επιστολές, τα γράμματα που έχω λάβει που μου λένε πηγαίνετε να βρείτε τον Τούσκ, η ψηφοφόρη μου, να του σφίξετε το χέρι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προσπάθειές του. Έχετε αναλάβει μια ευθύνη βαριά, μια ευθύνη να αντιμετωπίσετε την εκδοχή της εξόδου του Ρημανού Βασιλείου χωρί συμφωνία. Και αυτό ήταν μια βαριά ευθύνη για να αντιμετωπίσετε τα λάθη των συντηρητικών που έκαναν προχειροδουλειά και προκυρήσοντα ένα δημοψήφισμα για το οποίο δεν ήταν έτοιμοι. Η δουλειά του κυρίου Μπαρνιέ, του κυρίου Τούσκ, του κυρίου Γιουνκέρ πολιτικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο ήταν αυτοί που μα επιτρέπουν να συμμετάσχουμε στι 23 Μαου που διεξάγονται οι ευρωεκλογέ στη Βρετανία και του ευχαριστούμε γι' αυτό διατηρούμε την ελπίδα να μείνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην ε- Ηνωμένη Ευρώπη και είναι γενναίοι εκείνοι οι οποίοι βάζουν το μέλλον της χώρας μπροστά από τα μικροκομματικά συμφέροντα. Ήρθε η ώρα να ζητήσουμε να γίνει δημοψήφισμα το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε έως τις 31 Οκτωβρίου να έχει ληφθεί απόφαση ότι θα παραμείνουμε, ότι θα επικρατήσει το Remain. Ευχαριστώ, κύριος Ντάνς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ε, στα γαλλικά, να εκφράσω εκ μέρους του λαού της Ιρλανδίας ε, τη συμπόνια μας προς το λαό του Παρισιού για την καταστροφή της Πανηγίας των Παρισίων. Θα την ξαναχτίσουμε όλοι μαζί. Θέλω να τιμήσω και το θάρρος των πυροσβεστών. Συνάδελφοι, το Brexit είναι μια διαδικασία εν εξελίξη, την οποία αρνούνται αυτοί που κάθονται απέναντί μου, αρνούνται να κοιτάξουν ότι κάθε επιλογή που έχει μέσα της ένα Brexit, μια έξοδο, έχει αρνητικές συνέπειες τους. Είναι πολύ πιο εύκολο λοιπόν να κάθονται και να λένε «Α, μας προδώσατε» χωρίς όμως να πράττουν τίποτα, γιατί το Brexit δεν μπορεί να υλοποιηθεί όπως το υποσχέθηκαν. Ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε νέες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να δοθεί στο λαό η επιλογή να καταρρύψει όλους αυτούς που μιλούν για τα μονάχα Όλοι εμεί που είμαστε διατεθειμένοι από αυτήν εδώ την πλευρά να σταθούμε ε, στο πλευρό των Ευρωπαίων συμπολιτών μα και να χτίσουμε μαζί ένα κοινό μέλλον, είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε. Σα ευχαριστώ. Κύριε Χένκελ, ένα λεπτό. Πρώτη φορά πήγαμε το ποδήλατο από το Λουξεμβούργο μέσω Βελγίου στο Παρίσι ποδηλάτης για να επισκεφθώ την ε, Παναγία των Παρισίων και χτες την είδα να φλέγεται και δάκρυσα κυρίες και κύριοι. Είπατε κύριε Τούσκ ότι συμπονείτε το Παρίσι γιατί, είδατε, γιατί ξέρετε πως είχε καταστραφεί το Γκτάνσκ. Θα σας μιλήσω εγώ για την ε, ε Παναγία της Δρέσδης που χτίστηκε με την συνδρομή των Βρετανών των χτιστών που ήρθαν από το Κόβεντρι. Και θα πω ότι πρέπει να γίνει κοινό εγχείρημα για να ξαναχτιστεί η μεγάλη η Παναγία των Παρισιών, ο καθεδρικός ναός του Παρισιού. Πρέπει να είναι ένα κοινό εγχείρημα ευρωπαϊκό. Κύριε Τούσκ, είπατε επίσης ότι θα πρέπει και τα 28 κράτη να συμμετάσχουν. Την απάντηση πρέπει να τη δώσει το Λονδίνο βέβαια πια γιατί άκουσα και εσείς τι είπατε και ο κύριος Γιούνκερ. Αλλά κάτι πρέπει να πράξετε για να λάβετε τη σωστή απάντηση από το Λονδίνο. Αυτό πρέπει να πράξετε είναι να εξασφαλίσετε πως η Βρετανία θα παραμείνει και θα είναι μέλον, μέλος της προσπάθειας ανοικοδόμησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης της Παναγίας των Παρισίων για να μπορέσει να παραμείνει μέλος της ε, Ενωμένης Ευρώπης του Ρωμένου Βασίλειο. Κυρία Χιούμπνερ, για ένα λεπτό. Uh, uh, Ευχαριστώ. Πρόεδρε, συνάδελφοι για τους Ευρωπαίους ηγέτες η νέα προθεσμία για το Brexit ήταν δύσκολη απόφαση. Ε, τώρα η Βρετανική πλευρά θα πρέπει να χρησιμοποιήσει με επικοδημητικό τρόπο αυτό τον περαιτέρω χρόνο και σίγουρα δεν βασιζόμαστε στον κύριο Φαράζ. Είναι απογοητευτικό ότι την τελευταία εβδομάδα ακούσαμε σχόλια και είδαμε tweets ε, αντιευρωπαίων πολιτικών για το πώς θα σαμποτάρουν τη δουλειά μας στους επόμενους μήνες. Αυτή η πολιτικοί πρέπει να καταλάβουν ότι δεν πρόκειται να τους το επιτρέψουμε. Θα προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να αποτελεί την πηγή της σταθερότητας για, σε αυτήν την παράλογη διαδικασία του Brexit. Δυστυχώς από την Βρετανική πλευρά δεν υπάρχουν δεν υπάρχουν δείγματα ότι το, μια συμφωνία για το Brexit ε, θα επιτευχθεί. Το προβληματικό πρόβλημα δεν είναι το backstop, είναι το μέλλον. Και ίσως μια λύση να βρεθεί. Αυτό που χρειάζεται στη βρετανική πολιτική είναι το να οριστεί, να αποφασίσουν τι πραγματικά θα επιθυμούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σκέλη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να εκφράσω την ε, συμπάθειά μου και αυτή της Ιρλανδικής κυβέρνησης για την καταστροφή της ε, συμβολικής Παναγίας των Παρισίων. Τώρα, για το Brexit τόσο τραβάει, τόσο περισσότερο υποφέρει ο κόσμος και δυστυχώς αυτό ισχύει για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από το Brexit και για τους γεωργούς ε, που παίρνουν 100-200 ευρώ ε, λιγότερα αναζώ από ό,τι πέρυσι, ακριβώς λόγω αυτής της αβεβαιότητας του Brexit. Ελπίζω λοιπόν ο Τερέζα Μέι και ο Τζέρμι Κόρμπιν να φτάσουν σε μια συμφωνία, αλλά πολύ αμφιβάλλουμε. Εάν όχι, θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση για να αναβληθεί το Brexit επάπειρον. Θα πρέπει να ε, υπάρξει βεβαιότητα. Επίση, επηρεάζεται η περιφέρειά μου γιατί πρέπει να εκλεγούν πέντε μέλη στην Ευρωκοινοβούλιο ενώ τώρα φαίνεται πως θα εκλέξουμε μόνο τέσσερι. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε μόνο τους Βρετανούς γι' αυτό. Εγώ πριν από δύο χρόνια ζήτησα να μην δοθεί καμία έδρα μέχρι ότου να φύγουν οι Βρετανοί γιατί είχα πει ότι υπάρχει πιθανότητα να μην φύγουν μέχρι τις 29 Μαρτίου. Δυστυχώ βγήκα αληθινό. Ε, ε, εάν δεν ληφθεί απόφαση λοιπόν ε, για συμφωνία εξόδου, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ. Κάτσε διάει ο κύριο Ρανζέλ ένα λεπτό. Πρόεδρε, εγώ ήθελα να πω ότι με χαρά βλέπω πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έδειξαν ευελιξία με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είχαμε ζητήσει. Με χαρά βλέπω επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαθέσιμο για να οργανώσει ευρωεκλογέ και άρα ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα ο Βρετανικός λαός στο μέλλον να αποφασίσει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως θα ήθελα να είναι σαφές ότι αυτή η απόφαση εξακολουθεί να δημιουργεί μεγάλη αστάθεια για τους ανθρώπους, για τις εταιρείες και για τα κράτα ίδια. Ε, γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις εθνικές κυβερνήσεις να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους ώστε να ε, μπορέσουν να δώσουν ε, ε, βεβαιότητα στον κόσμο που υποφέρει λόγω αυτής της αναποφασιστικότητας του Βρετανικού Κοινοβουλίου και των αποφάσεών του. Κυρία Γκόμες, ένα λεπτό. Όλοι μας θρυνούμε για τη Γαλλία, για την ανθρωπότητα, γιατί η Παναγία των Παρισίων έχει χτιστεί από την ανθρωπότητα και η ανθρωπότητα θα την ξαναχτίσει. Θα ήθελα να πω πως λυπούμε πως το Συμβούλιο δεν έθεσε στην ημερήσια της για τη Βρετανία την υποχρέωση να ζητήσει ψήφο από τον λαό. Είναι ο δημοκρατικός τρόπος για να λυθεί αυτό το μπάχαλο, να αποφευχθεί προσπαθεί η Βρετανία να φύγει από την, την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω πως πλέον αυτό το μήνυμα θα πρέπει να σταλεί στο Βρετανικό λαό, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, στα Βρετανικά κόμματα από τους ηθήνοντες στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι επίσης θα αντιμετωπίσουμε και τα αίτια της αποξένωσης των πολιτών που, οποίο οποίο οφείλεται το Brexit αλλά και ε, δείχνει ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μεταρρυθμιστεί και να ξαναχτιστεί. Ευχαριστώ κυρία Μιράντα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή την Κυριακή πήγα στο Λονδίνο και μαζί με ένα σύλλογο Γαλλικιανών που είναι πολύ άριθμοι και ζουν στον Ηνωμένο Βασίλειο και υπάρχει αβεβαιότητα για την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, των υπηρεσιών και αβεβαιότητα επίσης για τα θέματα των ε, ε, ε, συνεπειών. Εργάζονται και ζουν στον Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι Ευρωπαίοι και Ευρωπαίες και δεν ξέρουν τι θα γίνει. Θέλω να πω επίσης, Πρόεδρε, και πρόεδρε Γιούνκερ για την πολιτική της ε, αλλίας ε, των υπηρεσιών με βάση τα όσα γίνονται εδώ, με το τέλος αυτής της θητείας, είναι δικιά μας υποχρέωση να δείξουμε ευελιξία για να μπορέσει ο κόσμος που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και που είναι Ευρωπαίοι να ε, ζήσει με μεγαλύτερη βεβαιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λόπες Ευχαριστώ. Πρόεδρε Γιούνκερ, η Ευρώπη πρέπει να περάσει σε άλλα θέματα. Πρέπει να συνεχίσει να βαδίζει προ τα μπρο και να επικεντρωθεί επιτέλου μετά από όλη αυτή την παγίδα του Brexit σε άλλα θέματα, για παράδειγμα, βλέπουμε πόσο θλιβόμεθα από την καταστροφή στο Νότρο Ντάμ. Στις 26 Μαου έχουμε μια υπαρξιακή σημασία εκλογική διαδικασία. Αλλά αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερε αβεβαιότητε για την σύνθεση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί έχει να κάνει με το αν θα συμμετάσχει όχι το Ηνωμένο Βασίλειο. Αναμένω λοιπόν να υπάρξει μία ε, απάντηση. Όχι μόνο δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία στη Βουλή των Κοινοτήτων, αλλά είναι πραγματικά απαράδεκτα ελαφρύ. Εδώ και 20 χρόνια καταδικάζουν ε, το ευρωπαϊκό εγχείρημα και επιτέλους περιμένω στις 26 Μαΐου οι φιλοευρωπαϊστές να συντρίψουν αποφασιστικά την δημαγωγία και την ευρωφαβία όχι μόνο στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπρέναν. Έχει περάσει ώρα και μας μένει λίγος χρόνος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομήθηκε με βάση την εμπειρία από τον εφιάλτη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πόλεμου και ένας οραματισμός λόγω αυτού του πολέμου μας οδήγησε στην κατάσταση όπου είμαστε σήμερα. Και συμφωνώ λοιπόν με τα σχόλια του Πρόεδρου Τάσκ. Χρειαζόμαστε ακόμη ονειροπόλου. Όπω είπε και ο Τζι Λόρεν, όλοι ονειρεύονται, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Όσοι ονειρεύονται τη νύχτα στο υποσυνείδητό του, ξυπνάνε τη μέρα για να βρουν ότι ήταν ματαιοδεξί όλα αυτά. Αλλά όσοι ονειρεύονται μέσα στη μέρα είναι επικίνδυνοι, γιατί μπορεί να επιχειρήσουν ε, με ανοιχτά μάτια να καταστήσουν πραγματικότητα τα όνειρά τους γιατί είναι αργά και μας μένει λίγος χρόνος. Πρόεδρε Τάσκ, σας καλώ να συνεχίσετε να ονειρεύεστε. Να ονειρεύεστε κι εσείς που είστε κατά της παραμονής, αλλά να μην ονειρεύεστε απλώς, να κάνετε πραγματικότητα τα όνειρά σας. Μπορούμε να παραμείνουμε. Θα παραμείνουμε. κύριος Χακμάρκ. Νομίζω ότι όλη η συζήτηση καταδεικνύει το εξής πόσο ισχυρή είναι η Ευρωπαϊκή Ενότητα. Τα προβλήματα στο Westminster δημιουργούνται από το ότι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει πολλά για μια κοινωνία και είναι δύσκολο να ε, διαραγούν αυτοί οι δεσμοί. Και είμαι ευγνώμων που ο κύριος Φάρατζ είναι αστείος, αλλά είναι απλώς αστείος. Ποτέ σοβαρά δεν έχετε συμβάλει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, στο άνοιγμα των αγορών στην Ευρώπη. Απλώς ήσασταν αστείος. Γιατί να σας φοβόμαστε. Προσπαθείτε να μας φοβήσετε λέγοντας ότι θα ξαναγυρίσουμε εδώ. Μα κοιτάξτε, είστε απλώς ο γελοτοποιός ε, στην αυλή. Αλλά δεν χρειάζεται να σας ακούμε. Αυτά που λέτε δεν έχουν καμία έννοια για την ενότητα ή για τους ε, λαούς της Ευρώπης. Είστε απλώς αστείος. Δεν σας φοβόμαστε και ελπίζω το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνει τη διαδικασία Catch the Eye. Να δώσω το λόγο τώρα στον πρόεδρο Γιούνκερ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παίρνω το λόγο ώστε να ευχαριστήσω τους βουλευτές τώρα από αυτά τα χρόνια που ερχόμαστε στο Στρασβούργο όλοι. Θα είμαι παρόν και στην έναρξη των εργασιών του Προσεχούς Κοινοβουλίου, αλλά θα μου λείψει ο καλός φίλος Έλμαρ Μπροκ όλα αυτά τα χρόνια, δουλέψαμε μαζί. Τσακωθήκαμε, συμφιλιωθήκαμε, γελάσαμε, πότε πότε κλάψαμε κιόλας. Ήταν τόσο ωραίο που συνεργαστήκαμε μαζί, Έλμαρ Μπροκ, και σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Γιουνκέρ, ο Πρόεδρος Τούσκ. Μια παρατήρηση μόνο, Πρόεδρε. Πολλές εβδομάδες τώρα. έχει προξενήσει έντονες αντιδράσεις στο ενδεχόμενο συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ευρωεκλογέ. Θέλω να υπενθυμίσω προς άπασα κατεύθυνση πως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει και δικαίωμα και υποχρέωση να λάβει μέρος στην εκλογική αυτή αναμέτρηση όσο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Επίσης, δεν δέχομαι να ε, εγκαθιδρυθεί δεύτερη κατηγο... δεύτερης κατηγορίας συμμετοχή κράτους μέλους. Αντιλαμβάνομαι ότι ορισμένα ε, κομματικά συμφέροντα μπορεί να επισκιάζουν ή να επιχειρούν να επισκιάσουν την νομιμότητα. Ο κύριος Φερχόφστατ ε, επικροτήθηκε ενθουσιοδός από τον κύριο Φαράς. Αυτό, κύριε Φερχόφστατ, θα έπρεπε για σας να αρκεί ως λόγος να αλλάξετε στάση και να διατυπώσετε με διαφορετικό τρόπο τα επιχειρήματά σας. Σας ευχαριστώ. Thank you. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση. Thank you, colleagues. You can continue the conversation συζητή σα μπορείτε να τις συνεχίσετε εκτό της αίθουσα τη ολομέλεια. Έχουμε άλλο θέμα τώρα. Παρακαλώ την Επίτροπο Τίσεν να έρθει στη θέση της ε, όσο περιμένουμε από τους ε, συναδέλφους που θα αποχωρήσουν όπως και τον κύριο Τούς, τον κύριο Μπαρνιέ, τον κύριο Γιουνκέρ και παρακαλώ οι χαριαντισμοί εκτός αιθούσης να συνεχιστούν. We Ενός ε, λεπτού διακοπή, μια και δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί η τάξη. Ενός λεπτού διακοπή. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ και πάλι να αποχωρήσετε εφόσον δεν σας ενδιαφέρει η επόμενη συζήτηση και δεν σκοπεύετε να συμμετάσχετε. Κύριε Κορμπέτ, κύριε Σμιθ, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσει η επόμενη συζήτηση. Παρακαλώ, επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Ενρίκε Κάλβετ Τσαμπών για τις διαφανείς, τους διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνω για 4,5 λεπτά το λόγο στον κύριο Κάλβετ Τσαμπών. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, ε, χαίρομαι που είστε μαζί μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Έχω τη τιμή να παρουσιάζω σήμερα την εργασία μιας ολόκληρης ομάδας, την οποία ευχαριστώ για τη συνεργασία που μου προσέφερα στη διάρκεια μηνών υπό χρονική πίεση, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και να προτείνουμε μια οδηγία που ε, θα αντικαταστήσει μια προηγούμενη οδηγία 28 ετών και που ε, προχωρά πολύ πιο πέρα. πολιτική σημασία αυτής της οδηγίας είναι πολύ μεγάλη σε αυτή την χρονική στιγμή. Αυτή η οδηγία εντάσσεται στην ανάπτυξη του κοινωνικού πυλώνα που ε, τούτη θητεία πάντοτε θα έχει, ε, θα, θα, θα, θεωρείται αυτή που προέταξε στο Γκέτεγμπουργκ πέρσι. Το πρώτο βήμα έγινε για την πραγματική πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στο κοινωνικό πυλώνα. Με αυτή την έννοια είναι μια οδηγία που επηρεάζει όλους τους εργαζόμενους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα όλους τους πολίτες που προετοιμάζονται για την αγορά εργασίας ή που εργάζονται ε, ήδη ε, ενώ ε, διεκδικούν αυτά τα δικαιώματα. Πρόκειται δηλαδή για εκατομμύρια κόσμο που καλείται να ψηφίσει μέσα σε ένα μήνα. Ε, και γι' αυτό και αποκτά και ιδιαίτερη σημασία ε, η έγκριση αυτής εδώ της οδηγίας εξισορρόπησης που ε, συμφωνήθηκε ανάμεσα σε όλες τις ε, συνιστώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ, σε αυτήν την οδηγία, τι γίνεται. Θεσπίζονται κάποια μήνυμα δικαιώματα που να είναι τα ίδια για όλους τους εργαζόμενους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δικαιώματα λοιπόν δεν θεσπίζει νόμους, δεν θεσπίζει μεθόδους, δεν θεσπίζει συγκεκριμένες εφαρμοστικές διατάξεις, γιατί αυτό θα εξαρτηθεί από τα κράτη-μέλη. Να είναι σαφές αυτό. Δεν υπάρχει καμιά επέμβαση, παρέμβαση στην αρχή της επικουρικότητας. Αυτό που θεσπίζει είναι δικαιώματα και ελάχιστες προδιαγραφές, ώστε στην Ευρώπη να μπορούμε να μιλάμε για για μια κοινωνική Ευρώπη όπου μπορεί κανείς να αναπτύξει την επαγγελματική του ζωή. Το περιεχόμενο είναι αυτό που γνωρίζουμε ε, καλύτερα, ε, δηλαδή δίνονται κάποια δικαιώματα ενημέρωσης ε, πολύ πολύ βελτιωμένα σε σχέση με την οδηγία του 91. Επίσης δικαιώματα μη κατάχρησης μη κατάχρηση ε, των ε, δοκιμαστικών περιόδων, ε, συγκεκριμένα δικαιώματα που είναι καθολικά για την Ευρώπη μόλις αυτή η οδηγία μεταγραφή και αποτελούν την αναφορά. Και επίσης σε μεγάλη σημασία έχει ότι καθορίζονται δικαιώματα ουσιαστικά τα οποία έχουν να κάνουν με όλες τις νέες μορφές ε, ε, ε, εργασίας, on-demand, platform, επισφαλής εργασίες. Όλοι αυτοί οι εργασόμενοι, δηλαδή που μέχρι τώρα ήταν σε ένα είδος <coughs> αοριστίας, τώρα θα καλύπτονται από αυτή την οδηγία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μπορεί να επικαλεστεί αυτή την οδηγία ώστε κανείς να μπορεί να καταχραστεί την απαραίτητη ευελιξία του χώρου εργασίας, του κόσμου της εργασίας. Επίσης είναι σημαντική αυτή η οδηγία σε επίπεδο, στο ισότιμο πεδίο για όλους. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει τονιστεί αρκετά. Δηλαδή εξασφαλίζει το ότι δεν θα επιβαρυνθεί η ποιότητα ζωής των εργαζομένων λόγω του κοινωνικού dumping αυτού του ε, φαντάσματος ε, που ε, υπήρχε μέχρι τώρα. Εμείς δηλαδή φτιάχνουμε την Ευρώπη και συγκεκριμένα την κοινωνική Ευρώπη. Ευχαριστώ όλους όσοι με βοήθησαν σε αυτή την εργασία. Σας ευχαριστώ. Κυρία Τάισεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριε Ευρωβουλευτέ, με μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ πριν την ψηφοφορία για αυτή την οδηγία, που είναι μία από τι βασικέ οδηγίε του Ευρωπαϊκού Πυλώνα το, για τα κοινωνικά δικαιώματα. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Καλβέτ Τσαμπόν που α, μπόρεσε να ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση αυτή τη οδηγία. Είχαμε χρονικού περιορισμού για να ολοκληρωθεί αυτή η οδηγία ε, από αυτήν τη θητεία γιατί, και χω, χω, χωρί την καλή για τη συνεργασία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα και χωρίς την ε, ακούραστη ε, προσπάθεια του εισηγητή για εξέβρεση συμβαστικών κειμένων στη διάρκεια της, εκπο... της... Ε, της διαπραγμάτευσης. Πρόκειται για επίτευγμα για την κοινωνική Ευρώπη, γιατί θα παρέχει στις 250 εκατομμύρια εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ευρώπη πιο διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας. Εξυγχρονίζεται το Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο και προσαρμόζεται στον νέο κόσμο της εργασίας. Όπως γνωρίζετε, ε, σήμερα ολοένα ε, και περισσότεροι εργαζόμενοι και κυρίως νέοι και εργαζόμενοι και κυρίως εργαζόμενες έχουν ε, πολύ πολύ ευέλικτες συμβάσεις εργασίας. Γι' αυτό και έπρεπε να βρεθεί σωστή ισορροπία, να εξασφαλίσουμε την προστασία για τους εργαζόμενους χωρίς να επιβαρύνουμε υπερβολικά τους εργοδότες και χωρίς να πνίξουμε την καινοτομία. Και αυτό ακριβώς κάναμε με την προτινόμενη οδηγία. Με τους νέους κανόνες λοιπόν θα εξασφαλίσουμε περισσότερη διαφάνεια πρώτο και κύριο. Όλοι οι εργαζόμενοι στην Ένωση θα πάρουν πληροφορίες για βασικές ε, συνθήκες εργασίας. Οι εργαζόμενοι θα γνωρίζουν εξ αρχής ε, Δηλαδή μέσα στην πρώτη του εβδομάδα ποια είναι τα βασικά του δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει πληροφορίες για την αμοιβή τους, για το χρόνο, πρόγραμμα εργασία τους, για τη διάρκεια της σύμβασής τους και χάρη στο Κοινοβούλιο και επιπλέον πληροφορίες για τους εργαζόμενους των ε, γραφείων προσωρινής απασχόλησης. Θα καλύπτονται ο, οι, οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι οικιακοί εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι με τις μηδενικές συμβάσεις και άλλου είδους ε, πρόθεσμοι εργαζόμενοι. Όμως δεν περιοριζόμαστε στην ενημέρωση, αλλά έχουμε και νέα ουσιαστικά δικαιώματα, όπως ας πούμε οι συγκεκριμένα στοιχεία για τις δοκιμαστικές περιόδους, η απαγόρευση αδικαιολόγητων ρητρών αποκλειστικότητας. Ε, επίσης, οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ποιες είναι οι χρονοθυρίδες που θα κληθούν να δουλέψουν και δικαίωμα σε αποζημίωση εάν διακοπεί σύμβαση εργασίας ε, χωρίς προειδοποίηση και τα λοιπά. Επίσης, για τις αρχές της υποχρεωτικής κατάρτισης θα πρέπει να είναι δωρεάν για τον εργαζόμενο και πάλι χάρη στο Κοινοβούλιο, θα πρέπει να μετρά ως χρόνος εργασίας η κατάρτιση. Άρα λοιπόν αυτά, αυτές είναι πιο δίκαιες συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους της Ένωσης. Ε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμοστούν σωστά οι κανόνες αυτοί θα δουλέψει η Κομισιόν σε συνεργασία με τι Εθνικέ Αρχέ ώστε να εξασφαλίσει τον τελικό στόχο συγκεκριμένα ε, δικαιώματα και για του ασφαλεί εργαζόμενου χωρί επιβάρηση για τι επιχειρήσει. Σα ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αρένα, ένα λεπτό από το πλευρά τη Επιτροπή Γυναικών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, σήμερα στην Ευρώπη πάνω από 4 εκατομμύρια εργαζόμενοι εργάζονται με συμβόλαια που τους καλύπτουν για λιγότερο από 8 ώρες τη βδομάδα και 1,6 εκατομμύρια έχουν ε, συμβόλαιο με ορισμένο χρόνο αλλά διάρκειας ε, για λιγότερο χρόνο και 6 εκατομμύρια ε, εργάζονται ακούσιο σε, για μερική εργασία και οι γυναίκες είναι πολύ πιο ευάλωτε σε τέτοιε συνθήκε και ενισχύονται αυτέ οι τάσει δυστυχώ. Οι θέσει εργασία που δημιουργήθηκαν μετά την κρίση του 2008 δυστυχώ συχνά, υπερβολικά συχνά, είναι επισφαλεί, κακοπληρωμένε, με ελάχιστη προστασία που δεν δίνουν καμία προοπτική στους εργαζόμενους οι οποίοι δεν μπορούν να δουν ποιο είναι το μεσοπρόθεσμο μέλλον τους δεν μπορούν να λάβουν ε, ένα τραπεζικό δάνειο δεν μπορούν να οργανώσουν τη ζωή τους το κείμενο που θα εγκρίνουμε σήμερα σίγουρα έχει στόχο να βελτιώσει την κατάστασή τους να τους εγγυηθεί καλύτερη προστασία και πάνω απ' όλα περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη ενημέρωση για τα συμβόλαια παντού στην Ευρώπη. Είναι σίγουρα πρόοδο, κύριε Επίτροπε και το είπατε. Ωστόσο, λυπάμαι, λυπάμαι που τα κράτη-μέλη αποκλείουν από την οδηγία τα συμβόλαια εργασία λιγότερο από 12 ώρε το μήνα και είναι απαράδεκτο που τα κράτη-μέλη δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στην απαγόρευση απλά και μόνο των συμβολίων μηδενικών ωρών θα έλεγα λοιπόν ότι ναι η Ευρώπη προτείνει μια πρόοδο είναι μια οδηγία ε, ελάχιστου ωφέλους αλλά τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι πιο φιλόδοξα για να προστατεύσουν του εργαζόμενού του. Αν θέλουμε οι εργαζόμενοι αυτοί, άνδρε και γυναίκε, να προσχωρήσουν στο ευρωπαϊκό όραμα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα οι πολιτικέ ομάδε. Ο κ. Ζωράτηκε, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι περήφανος για το αποτέλεσμα που έχετε ενώπιόν σας. Σίγουρα αυτό το αποτέλεσμα είναι ένα συμβασμό, ε, κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά εδώ στο σώμα μα. Αλλά οι καλοί συμβασμοί αποδεικνύονται από το ότι όλοι όσοι συμμετείχαν ε, σε ορισμένα σημεία, ένα-δύο, λένε ότι θα ήθελα κάτι περισσότερο ή θα ήθελα να τονίσω κάτι περισσότερο. Αλλά σε τελευταία ανάλυση και στην Επιτροπή, όπω υπόθηκε, υπήρξε ευρεία συνένεση και συνολικά πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση από πλευρά του ΕΛΚ. Λοιπόν, θέλω να τονίσω τα εξή. που ήταν πολύ σημαντικά και για μένα που ήμουν σκιώδης. Πρώτον, η νέα οδηγία υπάρχει περισσότερη προστασία ιδιαίτερα για τους ε, ε, επισφαλώς εργαζομένους. Και σωστά τόνισε η Επίτροπος ότι θα μειωθεί και η γραφειοκρατία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι όντω εκπροσωπούνται τα συμφέροντα και των μεν και των δε εργαζομένων και εργοδοτών. Επίση, κάτι άλλο πολύ σημαντικό για μένα και την ομάδα μου, τα καταφέραμε. Ο νομικό ορισμό του εργαζόμενου που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιηθεί στο κείμενο. Καταφέραμε ο ορισμό αυτό μάλλον να απαλληφθεί από το κείμενο και να ε, αποφασίζεται από τα κράτη-μέλη. Γιατί ένα ενιαίο ορισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα έφερνε περισσότερη νομική ασφάλεια, αλλά περισσότερη νομική αβεβαιότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η οδηγία θα βελτιώσει την κατάσταση των εργαζομένων και στη χώρα μου, που είναι περίφημο από πολλέ απόψει για την προστασία των εργαζομένων, αλλά παρόλα αυτά οι δεσμεύσει μέσω συλλογικών συμβάσεων αφορούν μόνο το 52% των εργαζομένων. Πολλοί εργαζόμενοι λοιπόν, θα, οι υπόλοιποι, θα ωφεληθούν από αυτή την οδηγία. Και κάτι που με εκνευρίζει στην προεκλογική εκστρατεία. Οι σοσιαλδημοκράτε, οι πράσινοι και οι αριστεροί λένε ότι η Ευρώπη είναι η Ευρώπη των τραπεζών και των επιχειρήσεων. Τότε πρέπει να του πω ότι αυτό το νομοθέτημα είναι σημαντικό τμήμα τη πρόθεση τη κοινωνική Ευρώπη και είμαι περήφανο γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου των Σοσιαλιστών Δημοκρατών, κύριο Λόπε, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα εγκρίνουμε αυτή την οδηγία για τι συνθήκε εργασία για να είναι προβλέψιμε και διαφανεί θα μας επιτρέψει το νομοθέτημα αυτό να προστατεύσουμε πάνω από 200 εκατομμύρια εργαζομένους στην Ευρώπη. Θα βελτιώσει τι συνθήκε εργασία των εργαζομένων που έχουν επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης με μη συνήθη και κακοπληρωμένα και με κακές συνθήκες συμβόλαια εργασίας. Θα τους δώσει εγγυήσει και ασφάλεια η οδηγία αυτή. Θα καλύψει και θα προστατεύσει του εργαζόμενου που εργάζονται σε ψηφιακέ πλατφόρμες. Σε πολλά κράτη-μέλη έχουν ανεπαρκή προστασία από κοινωνική πλευρά. Θα υπάρξουν και μέτρα για να καταπολεμηθούν οι, καταθρίσεις, οι καταχρήσεις των συμβουλέων ε, μηδενικών ορών ή αυτών που δουλεύουν με το κομμάτι. Πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα την Επίτροπο κυρία Τάισεν για την εργασία για το θέμα αυτό, την Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και επίσης ε, τους συναδέλφους στο Κοινοβούλιο και την Προεδρία του Συμβουλίου, τη Ρουμανική Προεδρία που έκανε ό,τι μπορούσε για να υποβληθεί σε, αυτό το τελευταίο, σε αυτή την τελευταία ολομέλεια ένα βασικό θέμα του πυλώνα των ε, κοινωνικών δικαιωμάτων. Δεν εγκρίνουμε απλώ κάποια μέτρα. Επιδεικνύουμε, καταδεικνύουμε μάλλον μια πορεία. Μια πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη. Μια χρήσιμη Ευρώπη. Προστατεύει που διεκδικεί την κοινωνική ψυχή της αποδεικνύουμε ότι η κοινωνική Ευρώπη δεν είναι απλώ ε, διακήρυξη προθέσεων. Καταλήγει σε συγκεκριμένα εργαλεία με συγκεκριμένε πιστώσει. Γιατί? Γιατί σήμερα η κοινωνική διάσταση του ευρωπαϊκού εγχειρήματο δεν είναι επίπτωση της ενοποίησης. Είναι προπόθεση για περαιτέρω ενοποίηση της Ευρώπη. Πρέπει να καταπολεμηθούν και να απαλληλθούν οι ανισότητε, Να προστατεύσουμε αυτούς τους οποίου θίγει η παγκοσμιοποίηση, να δώσουμε οικονομική ασφάλεια και προστασία στην αγορά εργασίας. Έτσι μόνο θα υπερασπιστούμε την ε, ευαίσθητη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Ευχαριστώ. κυρία Ένα Πρόεδρε, σε όλη μου την ε, θητεία εδώ στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Επασχόλησης υπερασπίστηκα ένα θεματολόγιο για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εδώ όμως δεν έχουμε καλύτερη νομοθέτηση με μια ε, σπουδή να ολοκληρωθεί το νομοθέτημα το χέτερο δυνατό ε, παρετούμαστε από τις προνομίες του Κοινοβουλίου δεν έχουμε σαφή ορισμό του αυτοαπασχολουμένου μόνο μέσα από μία αιτιολογική σκέψη ε, με πολύ λίγες λέξεις υπάρχει αυτή η αναφορά Πώ το δέχεται αυτό ο ΕΛΚ, πώς δέχεται η ομάδα των σοσιαλιστών για του ε, κυβερνήτε των αεροσκαφών τις αναφορέ που υπάρχουν για, την, ε, ε, για τον εργαζόμενο. Πρέπει να υπάρχει προστασία τη υγεία και τη ασφάλεια στο χώρο εργασία, σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση. Στον τριμερή όμως διάλογο έγινε η επιλογή να αποκλείεται αυτή η μεγαλη επιχειρηση στον τριμερη όμω διαλογο εγινε η επιλογη να αποκλειεται αυτη η διασταση των πυροσβεστών, των σωμάτων ασφαλείας, των δικαστών και εισαγγελέων και έτσι μπορούν τα κράτη-μέλη να αυτοεξαιρούνται, πράγμα το οποίο βεβαίως είναι εις βάρος του ίδιου του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της ΚΟΕ, η κυρία Λόπε Δεπερμαχώ για ένα λεπτό και 30 δεύτερα. Eh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του και ταυτόχρονα να εκφράσω τη λύπη μου που το, το Συμβούλιο για άλλη μια φορά ε, μπλοκάρισε οποιαδήποτε πρόοδο για τα δικαιώματα των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Εμεί θέλαμε να στηρίξουμε τους εργαζόμενους ε, που δουλεύουν με επισφαλείς συνθήκε και το κείμενο που θα εγκριθεί τους αφήνει σχεδόν χωρίς καμία προστασία. Αποκλείονται οι επίγουσες υπηρεσίες οι εργαζόμενοι στη θάλασσα, η οικιακή βοηθή, ε, οι ορισμένε συνθήκε, οι συμβάσει λιγότερο των 12 ωρών και ε, ε, μηνιαίω και πολλοί άλλοι εργαζόμενοι. Όπω λένε τα συνδικάτα, αυτά όλα αποτελούν διακρίσει και από κίνδυνο προηγούμενο σε σχέση με τα μήνυμα με δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εξ θα έπρεπε να είναι καθολικά. Εάν χαθεί ευκαιρία για οικοδόμηση μια κοινωνική Ευρώπη που ζητούν οι εργαζόμενοι. Αυτό που τίθεται επιτάπητος όμως είναι πιο βαθύ πρόβλημα και είναι η, ε, θεσμική, το θεσμικό μπλοκάρισμα όπου το Συμβούλιο, ε, τα κράτη-μέλη μπλοκάρουν διαρκώς τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι αυτό το οποίο ψηφίζουν οι, οι, πολίτες θέλετε να απομακρύνετε ακόμη περισσότερο τους πολίτες και την, ε, έτσι να επενθαρρύνετε την άνοδο της ακροδεξιάς. Ε, κυρία Λάμπερτ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, όπως και άλλοι ομιλητές εκ μέρους της ομάδας μου θα ήθελα να πω ότι πρόκειται και μια ευκαιρία χαμένη για εξυγχρονισμό της ε, οδηγίας. Εδώ βεβαίω θα μπορούσαμε να πούμε ότι καλωσορίζουμε μέτρα που έχουν να κάνουν με την καλύτερη ενημέρωση, πληροφόρηση, ε, αποζημίωση για ε, ακυρούμενη πρόσκληση σε εργασία, σε παροχή έργου μάλλον. Αλλά δεν ενημερώνεται σωστά ο εργαζόμενος και υπάρχουν πολλές εναλλακτικέ από διάφορα κράτη-μέλη, πράγμα το οποίο τελικά υπονομεύει την έννοια της ασφάλειας δικαίου και υπάρχει ζήτημα σε σχέση με την πρόθεση κρατών μελών να καλύψουν ως το, το πεδίο εφαρμογής λιγότερους ακόμη εργαζομένους και όχι μόνο αυτά που αναφέρθηκαν νωρίτερα, δημόσιους υπαλλήλους, ε, υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης, ε, εργαζόμενους ε, στην στα οικιακά σε έναν βαθμό, αλλά και την, ανάγκη, και την ανάγκη που δεν επιβάλλεται στα κράτη-μέλη να επενδύσουν σε καλές δημόσιες υπηρεσίες και να προβάλλουν την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης. Επίσης υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν σε διαφορετικές θέσεις εργασίας ή έχουν ε, συμβάσεις ε, ολίγων ωρών, συμβάσει έργο λίγων ωρών. Έτσι λοιπόν... Ε, οπωσδήποτε θα έπρεπε να έχει γίνει δεκτή η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσε το Συμβούλιο να το έχει πράξει και να δώσει περισσότερη σάρκα και οστά στην ουσία τη ε, απασχόληση. Αλλά αυτό που δίνει με το ένα χέρι το Συμβούλιο το παίρνει με το άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μελά. Δύο λεπτά. Ενφ. Πρόεδρε, ευχαριστώ προβλέψιμες και διασφανείς συνθήκε εργασία σταθερότητα στις συμβάσει ε, έργου για την καλύτερη αποζημίωση και αμοιβή των εργαζομένων είναι στόχος. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε μια γρήγορη... Πρέπει να αντιμετωπίσουν μάλλον οι εργαζόμενοι αλλά και οι εργοδότες μια εξέλιξη και μια επανάσταση ουσιαστικά της ε, αγοράς εργασίας με 20% θέσεων εργασίας που έχουν να κάνουν με, τις... με επισφάλεια, που είναι επισφαλιστέ εργασία. εργασίας. Νέες πρακτικές που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να προβλέψουμε όμως και να προλάβουμε και την κατάχρηση στις... στους εργαζομένους στα οικιακά σε πολύ περιορισμένη διάρκεια εργασίας εργασία, σε εργασία που σχετίζεται με τις ψηφιακές, ε, ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά και την εργασία που σχετίζεται με τις επιταγές, ε, τις οριές. Ε, αμοιβή. Ε, εκ μέρου τη ομάδα μου, λοιπόν, ε, έχω καταθέσει προτάσει, έχω υποστηρίξει κάποιε από τι συγκεκριμένε προτάσει του εισηγητή, θεωρώντα ότι είναι απαραίτητο να προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτω του πόσο επισφαλή είναι η θέση εργασία. Μην ξεχνάμε ότι η φτωχοποίηση γενικεύεται, η Ευρώπη με τις πολιτικές της. Ε, βεβαίως είναι υπεύθυνη γι' αυτό, είναι υπεύθυνη για, τους, ε, για τις ε, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδων αυτών των μικροθέσεων εργασίας, των mini jobs και είμαστε αντίθετοι σε αυτά τα μοντέλα τα οποία πρέπει προσπαθούν κάποιοι να μας επιβάλλουμε. Βεβαίως όμως έχοντας αυτό υπόψη ξέρω ταυτόχρονα ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα γιατί είναι υπαρκτά. Είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ε, παρισφρήσει στα παιδιά, αρμοδιότητα και κυριαρχία των κρατών μελών. Εμεί αγωνιζόμαστε ω ομάδα για ασφαλεί θέσει εργασία, για σίγουρες θέσει εργασία, με συνθήκε υγεία, ασφάλεια και ε, οικογενειακού βίου. Ευχαριστώ πολύ. Μπάλτσο, ένα λεπτό. Πρόεδρε. Το Νοέμβριο του 2017 στο Γκέτεμπορκ ε, εξασφαλίστηκε συμφωνία για τον κοινωνικό πυλώνα ο οποίος πανηγυρικά ανακηρύχθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που υπέγραψαν τη σχετική διακήρυξη. Εδώ υπάρχει μια προσπάθεια να αναπτυχθεί αυτός ο κοινωνικός πυλώνας. Έχει, έχει λεπτομερείς κανόνες για την, για την κοινή αγορά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο πια έχει έρθει η ώρα να αρχίσει και η δουλειά για τους εργαζομένους με την εισαγωγή ελάχιστων προδιαγραφών. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που δεν έχουν συγκεκριμένη ορισμένη, σύμβαση ορισμένου χρόνου απασχόλησης, ε, η Ουγγαρία έχει δει την έγκριση ενός συστήματος απασχόλησης από τις ε, κυβερνητικές δυνάμεις που οδηγεί σε συνθήκες σύγχρονης ε, δουλείας και που καταρρύπτει το κοινωνικό μοντέλο ε, με την εκμετάλλευση του εργαζομένου, με τις νέες ευέλικτες μορφές εργασίας που καταδικάζουμε. Ευχαριστώ. Κύριος Κάζα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του. Ε, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει αλλάξει η φύση της εργασίας. Πρέπει λοιπόν και εμείς να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να ενημερώσει τους κανόνες, να εξυγχρονίσει το πλαίσιο. Είναι ένα μικρό βήμα, αλλά άλλο ένα μικρό βήμα για μια πιο κοινωνική Ευρώπη για αυτό το θέμα. Την τελευταία πενταετία έχουμε εργαστεί ιδιαίτερα και ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο Τίσεν που έχει κάνει πολλά καλά και το, αλλά και τον πρόεδρο Γιούνκερ. Μαζί με τους συναδέλφους εδώ στο Σώμα και ιδιαίτερα την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα γίνει πιο κοινωνική από ό,τι ήταν ε, στο παρελθόν. Και είναι αναγκαίο αυτό το νομοθέτημα γιατί σήμερα οι θέσει εργασία γίνονται όλο και πιο ψηφιακέ, αλλάζουν τα συμβόλαια και είναι πολύ διαφορετικά. Η εργασία αποκτά ε, διάφορα μη ε, συνηθισμένα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, αυτά τα συμβόλαια με το κομμάτι μηδενικών ορών ε, εξαπλώνονται όλο και περισσότερο και αυτή η οδηγία προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες καταστάσεις. Γι' αυτό χρειαζόμαστε να προστατεύσουμε περισσότερο τους εργαζόμενούς μας ιδιαίτερα τους εργαζόμενους στις ψηφιακές πλατφόρμες. Για μια φορά ευχαριστώ όσους συμμετείχαν. Χάρη στην προσπάθειά τους έχουμε αυτό το πολύ καλό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Δεν βλέπω τον κύριο Ζημών. Ο κύριος Οκ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε η οδηγία για τις ε, διαφανείς και με συνθήκες εργασίες είναι ενδιαφέρον θέμα. Στόχος της είναι να δημιουργήσει περισσότερη ασφάλεια αλλά και περισσότερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις θέσεις εργασίας. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση επίσης να απολαμβάνουν ορισμένων, ε, ενός ορισμένου επίπεδου βεβαιότητας. Αυτό πρέπει να ισχύει και σε όσους εργάζονται σε μη συνήθεις ε, και επισφαλείς ε, μορφές εργασίας. Αυτό θα βοηθήσει και τις επιχειρήσεις, γιατί οι εργαζόμενοι θα είναι πιο αποδοτικοί. Πρέπει λοιπόν να ικανοποιήσουμε και τους μεν και τους δε. Και αυτοί είναι οι στόχοι. Αλλά το κείμενο αυτό όντω τους επιτυγχάνει. Όχι εντελώ. Πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα και περισσότερη προσαρμοστικότητα. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση τη αγορά-εργασία. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε υπερβολική γραφειοκρατία μικρομεσαίε. Ευχαριστώ πολύ. Ουρτασούν ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρά την καλή εργασία του Κοινοβουλίου, για την οποία ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ όσου συμμετείχαν, το Συμβούλιο αποδυνάμωσε ε, σε μία κλειδιά αυτού του θεμελιώδους νομοθετήματος για την κοινωνική Ευρώπη. Χάσαμε τον ορισμό που να τα περιλαμβάνει όλα τι σημαίνει εργαζόμενος και το τελικό κείμενο δίνει μεγάλες δυνατότητες στα κράτη-μέλη για να χορηγούν εξαιρέσει στου εργαζόμενου που εργάζονται λιγότερο από 12 ώρες το μήνα και για ένα μακρύ κατάλογο επαγγελμάτων όπω καταγγέλουν τα συνδικάτα. Επίση, χρειάζεται γραπτό συμβόλαιο από την 7η μέρα και μετά. Αυτό σημαίνει ότι όσοι εργάζονται στη μαύρη θα εργάζονται μόνο 6 μέρε για να μην φοβηθούν τον επιθεωτή εργασία. Όπω ε, υπόθηκε, δεν απαγορεύονται, τα ξεδιάτροπα συμβόλαια μηδέν ωρών που θίγουν πολλού συμπολίτε μα. Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται σε επιφελεί εργασίες και δεν προστατεύονται επαρκώ. Η κοινωνική Ευρώπη χρειάζεται φιλοδοξία και όχι αυτά τα παζάρια στα οποία έχουμε συνηθίσει στο Συμβούλιο. Παρά τα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. ένα λεπτό. οδηγία γνωστοποίησης των όρων εργασίας στους εργαζόμενους όχι απλά κοροϊδία περί δίθεν κοινωνικής ευρώπης μέσα από το ελάχιστο νομιμοποιείται το χειρότερο δεν δίνεται δικαιώματα στον εργαζόμενο στους εργοδότες δίνεται αρκεί να ενημερώνουν βέβαια πασάροντας ένα ραβασάκι για τους όρους της εργασιακής ζούγκλας. νομιμοποιείται τις πιο βάρβαρες μορφές εργασίας όπως συμβάσει μηδενικών ωρών προστατεύοντας την ευελιξία των εργοδοτών όπως λέτε αποκλείεται χιλιάδες οικιακούς βοηθούς ναυτεργάτες και άλλους ακόμα και από αυτό. ιδού ο ευρωπαϊκός κοινωνικός πυλώνας που ψήφισαν σύριζα νέα δημοκρατία και πασόκ. η ευρωπαϊκή ένωση μόνο προς το χειρότερο αλλάζει γιατί δεν αλλάζουν τα μονοπόλια που την έστησαν. στις ερχόμενες ευρωεκλογέ η λαϊκή δυσαρέσκεια να μην εγκλωβιστεί σε υποσχέσεις βελτίωσή τη σοσιαλδημοκρατών τύπου σύριζα και άλλων ούτε στον ευρωσκεπτικιστικό εθνικισμό για τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών κάθε κράτους ξεχωριστά να βρει ο λαό το δικό του δρόμο τον ταξικό ενίσχυση όσων στοχεύουν στην καρδιά του θηρίου τον καπιταλισμό την ευρωπαϊκή του ένωση τα μονοπόλια σε κάθε κράτος ενίσχυση του κομμουνιστικού κόμματο ελλάδας. κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Κομισιόν ήταν πολύ συνεπής. Σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ Επίτροπε Τάισεν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων που γίνεται πραγματικότητα. Αυτή η νέα οδηγία είναι σημαντική για όλους, αλλά ιδίως για αυτούς που εργάζονται επί τη βάση ε, άτυπων ε, συμβάσεων εργασίας για διάφορες πλατφόρμες ίντερνετ, μηδενικές ε, συμβάσεις μηδενικών ορών κτλ. 50% των νέων ε, θέσεων επασχόλησης είναι δεν είναι ε, χαρακτηριστικές. Ε, δεν καλύπτονται οι άνθρωποι αυτοί από την ισχύουσα οδηγία για τις γραπτές δηλώσεις. Γι' αυτό αυτό το νέο έγγραφο είναι πολύ σημαντικό, γιατί δίνει στους εργαζόμενους περισσότερα δικαιώματα, περισσότερη ενημέρωση και πιο σύντομα. Και περισσότερες λεπτομέρειες θα πρέπει να τους δίνονται. Αλλά πάνω απ' όλα η οδηγία αυτή θα καλύψει ε, μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων με βάση ε, ε, αυτούς που τις νέες μορφές εργασίας. Μόνο αυτοί που δουλεύουν λιγότερο από 12 ώρες το μήνα δεν καλύπτονται. Ε, πρέπει, είναι ιδιαίτερα καλή αυτή η οδηγία για τις γυναίκες. Πρέπει με, με έξυπνο τρόπο να καλύψουμε την ασφάλεια και την ευελιξία. Ευχαριστώ, η κυρία Μπένι Φέη. Ο κύριος Μπένι Φέη, συγγνώμη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο αριθμό των Ευρωπαίων πολιτών που εργάζονται σε επισφαλεί θέσει εργασία αυξάνεται διαρκώ και στην Ιταλία, βέβαια, βλέπουμε ότι επεκτείνονται διαρκώ και οι τομεί τη οικονομία με τι ψηφιακέ πλατφόρμε και αυτό που υποφέρει περισσότερο είναι ο νέο, είναι η γυναίκα εργαζόμενη. Πάνω απ' όλα με τι ατυπικέ μορφέ εργασία που, επε... που εξελίσσονται και συχνά είναι είτε χαρακτηρίζεται είτε αυτόνομη απασχόληση είτε μηδενικών όρων σύμβαση. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη διαφάνεια αλλά και ασφάλεια ως προς συνθήκες εργασίας αυτών των εργαζομένων με τα δικαιώματά τους τα οποία θα πρέπει για εκατομμύρια των εργαζομένων εξασφαλιστών. Πρέπει να κάνουμε περισσότερο. Εμείς ως σοσιαλιστές δημοκράτες θα συνεχίσουμε να απαιτούμε μία οδηγία για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζομένους που είναι σε εξαρτημένη σχέση και πρέπει να συνεχίσουμε έναν αγώνα ουσιαστικό προβάλλοντας τα δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως κάναμε στην από τρία χρόνια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αλλάξουμε πλέον την πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρικε, ένα λεπτό. Πρόεδρε, αξιότιμη επίτροπε. Η μερική απασχόληση συνήθως αναλαμβάνουν περισσότερο οι γυναίκες και δι οι μητέρες. Εδώ ακριβώς το χώρο της απασχόλησης θα έπρεπε να έχει εξασφαλιστεί η συμμετοχή των γυναικών, η αναγνώριση της ε, δουλειάς που κάνουν στην ανατροφή, στη μέρημνα για τα παιδιά, στη φροντίδα, σαν να ήταν παιδική σταθμή ή βρεφονικπιακή σταθμή που πληρώνουμε, θα έπρεπε να αμείβεται και η απασχόληση αυτή της γυναίκας. Ωστόσο, και αυτό θα βοηθούσε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν το κενό στην κάλυψη των σταξιδοτικών αναγκών για την επόμενη γενιά που ήδη διαφαίνονται. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Η Ουγγαρία θα μπορούσε μάλιστα να είναι υπόδειγμα στην περίπτωση αυτή όσον αφορά πάνω απ' όλα την αναγνώριση της προσφοράς των γονέων. Στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο λοιπόν ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο αυτό γιατί είναι ένα γιγάντιο έργο, ένα Ηράκλειο έργο μπροστά μα. Ευχαριστώ κυρία Σόιτροβα για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πρέπει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ε, εσωτερικής αγοράς. Η αγορά εργασίας μεταλλάσσεται ταχύτατα, είναι όλο και πιο ευέλικτες οι μορφές εργασίας που ε, προβάλλονται δεν τις θεωρώ εγώ και δεν τις χαρακτηρίζω επισφαλείς. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι η ευέλικτη απασχόληση μπορεί ή πρέπει αναγκαστικά να οδηγεί σε εκμετάλλευση του εργαζομένου. Υπάρχουν εργαζόμενοι που προτιμούν τις ευέλικτες συνθήκες εργασίας. Βεβαίως θα πρέπει αυτή η δουλειά να έχει μια προβλεψιμότητα αλλά και ασφάλεια για τον εργαζόμενο και υπ' αυτή την έννοια υποστηρίζω την οδηγία και τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί. Σας ευχαριστώ κύριε Ισηγητά, ευχαριστώ κύριε επίτροπε.